την κοινοβουλευτική θητεία, απαντώντα σε όλου αυτού του πολίτε που τα τελευταία πέντε χρόνια έρχονται σε επαφή μαζί μα. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε, κυρία Ματσόνη. Μία από τις ε, ιδιαιτερότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι κανένας δεν έχει την πλειοψηφία. Ήδη υπάρχει μια σταθερή πλειοψηφία. Ο σχετισμός δυνάμεων αλλάζει ανάλογα με την έκθεση και το συγκεκριμένο θέμα. Και δεν ξέρουμε ακόμη την έκβαση των επόμενων ευρωεκλογών. Γι' αυτό και καλό θα ήταν να κρατήσουμε αυτό το πνεύμα συνεργασίας που χαρακτηρίζει τις συζητήσεις μας. Η συζήτηση ολοκληρώνεται, θα ψηφίσουμε αργότερα στις 12. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, την έκθεση του κυρίου Παναγιώτοφ ε, που αφορά την πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τραποποίηση τη οδηγία σχετικά με τι ηλεκτρικέ στήρες και του ισορρευτέ για τα απόβλητα ηλεκτρικών στυλών που περιέχουν κάδμιο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από χρονοβόρε διαπραγματεύσει μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταλήξαμε τελικά σε μία φιλόδοξη αλλά ρεαλιστική συμβαστική λύση σε ό,τι αφορά την οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες και τους σωρευτές που περιλαμβάνουν κάδμιο. Ε, θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα στοιχεία σε σχέση με την τελική συμφωνία στην οποία καταλήξαμε. Στη διαπραγματεύση του τριμερούς διαλόγου καταλήξαμε σε μια συμβαστική λύση για την εξαίρεση τέτοιων ηλεκτρικών στυλών με κάδμιο σε ε, ηλεκτρικά, ηλεκτρικό εξοπλισμό που ε, ε, ολοκληρώνεται στα 2016. Ελπίζω ότι με τη συμφωνία αυτή θα υπερψηφίσουμε την συμβαστική λύση και θα βελτιώσουμε την τρέχουσα νομοθεσία γεφυρώνοντας σημαντικά κενά που υπήρχαν στην οδηγία. Στόχος των, της διάταξης αυτής είναι να επιτρέψουμε ολιγοδάπανη μετάβαση όλων στην ε, αλυσίδα παραγωγής και να βελτιώσουμε και το περιβάλλον και την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Πιστεύω ότι η τελική συμφωνία στην οποία καταλήξαμε δίνει ένα σαφές και στεναρό μήνυμα σε όλους για την απαγόρευση ε, του καδμίου στις ηλεκτρικές στήλες. Δεύτερο στοιχείο της πρώτης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η συμπερίληψη και του υδραργύρου στη συζήτηση για τις ε, ηλεκτρονικές μπαταρίες ό,τι φορά ιδιαίτερα τα στοιχεία κουμπιά που περιέχουν ε, υδράργυρο. Ε, χαίρομαι που οι συνάδελφοι της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, υποστήριξαν την έκθεσή μου για τα στοιχεία κουμπιών που περιέχουν υδράργυρο θα απαγορευτούν από την αγορά από το 2015. Είναι πολύ σημαντικό γιατί 5.000 ε, ε, μονάδες υδραργύρου θα αποφευθούν να ε, φτάσουν στο περιβάλλον. Και χαίρομαι γιατί με τη συμφωνία αυτή έχουμε μια πολύ φιλόδοξη συμφωνία για την οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες και τις σωρευτές και έτσι θα μπορέσουμε να ε, καινοτομήσουμε σε νέες τεχνολογίες και νέα υλικά και ταυτόχρονα θα δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα σε ό,τι αφορά το κάτμιο και το υδράργυρο και την ε, απέτησή μας να μην χρησιμοποιούνται πια και να μην μολύνουν το περιβάλλον. Ευχαριστώ θερμά και τους ε, σκιώδη γιατί χωρίς τη δική τους ε, αμέριστη υποστήριξη δεν θα μπορούσα να καταλήξω στο έργο. Μπόκοβιτς, Λιουτέρ, Μιροσλαφ Στάλκα Ευχαριστώ θερμά όλους αυτούς τους συναδέλφους για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε. Και θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν τη συμφωνία στην οποία κατέληξε Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο λόγο έχει ο κύριος Επίτροπος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή, τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτοφ και τους ε, συναδέλφους του για την επεξεργασία της πρότασης ε, της Κομισιόν να απαγορευτεί η χρήση καδμίου σε μπαταρίες ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων. Έχουμε λοιπόν τη σχετική μελέτη και το τελικό αποτέλεσμα είναι νομίζω καλά νέα για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η απαγόρευση υδραργύρου και καδμίου είναι άλλο ένα βήμα για να δημιουργήσουμε ένα μη τοξικό περιβάλλον, κάτι το οποίο στήριξε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος ε, δράσης για το περιβάλλον. Θα υπάρξει έτσι καινοτομία για να αναζητηθούν πιο ασφαλείς ε, εναλλακτικές. Η πρόβλεψη για την ε, αφαιρεσιμότητα των ε, μπαταριών σημαίνει πως θα μειωθούν τα απορρίμματα και θα αυξηθεί και η ανακύκλωση. Η Κομισιόν έχει καταστήσει σαφές πως υποστηρίζουμε το αποτέλεσμα όσον αφορά την ουσία σε κάποια διαδικαστικά ζητήματα οι αλλαγές που έγιναν στην πρόταση της Κομισιόν ε, μας αναγκάζουν να κάνουμε τρεις ανακοινώσεις. Αφορούν την χρήση της ρήτρα μη γνωμοδότησης για τις πράξεις εξοδότησης, συμμετοχή των ενδιαφερομένων και την δημοσίευση μιας ενοποιημένης οδηγίας. Θα δώσουμε τις οδηγίες αυτές στην γραμματεία για τα πρακτικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Κούκοβιτς, κυρία Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η αλλαγή, η τροποποίηση αυτή τη οδηγία για τι ηλεκτρικέ στήλε πραγματικά παρέχει πάρα πολλέ βελτιώσει για το περιβάλλον, για του τελικού χρήστε, για του καταναλωτέ και δημιουργεί μια προστιθέμενη αξία για τι καινοτόμε επιχειρήσει. Γνωρίζουμε πραγματικά πόσο πολύ εξαρτώνται η ζωή μα από τι ηλεκτρικέ στήλε. Οι ηλεκτρικέ στήλε ουσιαστικά παρέχουν ενέργεια την οποία δεν βλέπουμε. Χάρη στι ηλεκτρικέ στήλε, χάρη στι μπαταρίε μπορούμε να υποφεληθούμε από όλε τι σύγχρονε τεχνολογίε και χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο, όπω το γνωρίζετε, ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία. Παράλληλα όμω αυτέ οι ηλεκτρικέ στήλε βάλουν κατά του περιβάλλοντο και κατά τη ίδια τη ανθρώπινη υγεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να τροποποιηθεί, να ανανεωθεί, ή να αναθεωρηθεί, με συγχωρείτε, η νέα αυτή οδηγία ακριβώ επειδή έχουμε νέα επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά την περιβαλλοντική επίπτωση που έχουν ηλεκτρικέ στήλε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μία απαγόρευση για τι ηλεκτρικές στήλε νικελίου καδμίου. 16 εκατομμύρια τέτοιες ηλεκτρικές στήλες πολλούνται σε αιτήσια βάση, αλλά ένα 40% μόνο των ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων, των ηλεκτρικών μάλλον εργαλείων είναι ασύρματα. Ξέρετε ότι το κάδμιο έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία. Διαρρέει στο περιβάλλον, ακριβώς επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτε οι οποίοι δεν φροντίζουν να κάνουν σωστή διαλογή των αποβλήτων ηλεκτρικών στυλών. Εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλύσαμε την πρόταση αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ουσιαστικά την υποστηρίζουμε. Θεωρούμε ότι η τροποποίηση τη οδηγία και προστατεύει του καταναλωτέ και δίνει και μια μεταβατική περίοδο προκειμένου οι καταναλωτέ να καταφέρουν να προσαρμοστούν στο νέο νομικό καθεστώ. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλέ στήλε νικελίου καδμίου που υπάρχουν σε όλα τα νοικοκυριά ουσιαστικά, σε πάρα πολλέ συσκευέ. Υπάρχουν όμω πλέον νέες συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούν στήλες ιόντων λιθίου, οι οποίες όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται στα σύρματα ηλεκτρικά εργαλεία. Σύμφωνα με τη νέα οδηγία επίσης θα έχουμε και μία απαγόρευση στη χρησιμοποίηση υδραργύρου στα στοιχεία κουμπιά. Η, τα στοιχεία αυτά κουμπιά μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, ιδίω για την υγεία των παιδιών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Παναγιώτοφ τη χάρη στην τεχνική του πυρογνωμοσύνη στα ζητήματα αυτά καταφέραμε πραγματικά να βελτιώσουμε πάρα πολύ το κείμενο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εξ ονόματος ομάδας των Σοσιαλιστών, η κυρία Σάρμπου. μισή λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το 2006 είχαμε την οδηγία αυτή και τελικά εμ, επιτράπηκε εξαίρεση για ορισμένα χρόνια, αλλά μην ξεχνάμε ότι το κάδμιο είναι τοξικό και προκαλεί καρκίνο και καρδιακές ασθένειες σε πολλές περιπτώσεις. Ο υδράτυρος επίσης είναι πολύ επικίνδυνος και είναι γνωστά τα αποτέλεσματά του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει την ευθύνη να προστατεύσει όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και τη δημόσια υγεία και οι κίνδυνοι σχετικά με την ε, υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον μερικές φορές ε, έρχονται σε αντιπαράθεση με τα συμφέροντα της βιομηχανίας. Θα πρέπει λοιπόν ο κανονισμός μας ε, να είναι ισορροπημένος και θεωρώ ότι βρήκαμε τελικά την επιθυμητή ισορροπία γιατί με τη μείωση αυτών των τοξικών ουσιών στη χρήση, στις, στις ηλεκτρικές στήλες που χρησιμοποιούνται στα νοικοκυριά και στα σύρματα ηλεκτρικά εργαλεία θα περιορίσουμε την έκθεση των συμπολιτών μας σε τέτοιες τοξικές ουσίες, ενώ ταυτόχρονα θα ενθαρρύνουμε τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών πιο φιλικών προς το περιβάλλον και τη χρήση και καινοτόμων υλικών. Τελικά η συμφωνία αυτή είναι πολύ επιτυχής γιατί όχι μόνο θα μειώσει τη μόλις στο περιβάλλον αλλά και το κίνδυνο στην ανθρώπινη υγεία. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που το Συμβούλιο δέχτηκε την πρόταση του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό των οικιακών συσκευών και των ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων προκειμένου να γίνει εύκολη η αλλαγή των ηλεκτρικών στυλών. Αυτή τη στιγμή μεγάλος αριθμός ε, συσκευών ε, δεν έχει καλό σύστημα για την αλλαγή των μπαταριών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξανόματος τον Πρασίνο, ο κύριος Σλίτερ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το κάδμιο και ο υδράργυρος είναι δύο τοξικά βαρέα μέταλλα και τώρα επιτέλους αυτό το οποίο είχαμε επιτύχει το 2006 θα γίνει πραγματικότητα. Θα έχουμε πλήρη απαγόρευση αυτών των ουσιών στις ε, μπαταρίες σε μορφή κουμπιών σε 21 μήνες. Θετικό αυτό και μετά μέχρι το τέλος του 2016 θα καταργηθούν σταδιακά και οι εξαιρεσει ε, που είχαν εισαχθεί λόγω των επιχειρημάτων που προέβαλαν διάφοροι λομπίστες. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παναγιώτοφ, εξαιρετική η δουλειά του και αυτό σημαίνει πως ε, όλοι μπορέσαμε να συμφωνήσουμε. Επίσης είμαι υπερήφανος για το ότι επιτέλους ε, πραγματοποιήθηκε αυτό το οποίο ζητούσαμε την ε, τελευταία φορά. Ότι δηλαδή θα, υπάρχει, θα είναι υποχρεωτική η ανακύκλωση των μπαταριών και βεβαίως και η ευκολία στην αλλαγή τους. Γιατί αν αλλάξει κανείς την μπαταρία σε ένα προϊόν Apple χρειάζεται 110 ευρώ. Πρέπει να υπάρξει και εκεί ανταγωνισμός. Επίσης να σας υπενθυμίσω πως ήδη το 2009 έπρεπε να ε, έχει υπάρξει ένα σηματάκι για τις μπαταρίες μίας χρήσης και ακόμη το περιμένουμε. Όταν αγοράζει κανείς τις μπαταρίες πρέπει να γράψει το πακέτο τι περιέχει. όπως όταν πάμε στο βεζινάδικο, έτσι. Αναγράφεται πάνω και το προϊόν και η ποσότητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκολσον για τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζω την ε, τελική αυτή συμφωνία στην οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες, αν και εγώ θα ήθελα μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο. Η 31η Δεκεμβρίου 2016 είναι αποδεκτή αν δούμε πως Ήδη υπάρχουν περιορισμοί για την θέση σε εμπορία και βέβαια θα επιτραπεί να εξαντληθούν τα αποθέματα που υπάρχουν ήδη στα καταστήματα. Αυτό πάρα πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η απόφαση απαγόρευσης ε, του υδραργύρου στις στήλες με μορφή κουμπιού είναι πάρα πολύ σημαντική και συμμορφωνόμαστε έτσι και με την ε, σύμβαση του ΟΗΕ για την απαγόρευση της χρήσης του υδραργύρου μέχρι το 2020. Και βεβαίως θα πρέπει να δοθεί χρόνο σε επιχειρήσεις να προσαρμοστούν η ε, εξαίρεση που υπάρχει είναι πάρα πολύ σημαντική και την ε, υποστηρίζω, οπότε μπορούμε να στηρίξουμε την θέση αυτής της οδηγίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πάσκα έχει το λόγο για την Ευρώπη της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Γνωρίζουμε όλοι ότι η παραγωγή και η χρήση ηλεκτρικών στυλών και συσσωρευτών με κάδμιο είναι προβληματική όσον αφορά το περιβάλλον, τις πολύ αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ξέρετε ότι το κάδμιο μπορεί να περάσει ακόμα και στον ανθρώπινο οργανισμό, είναι πάρα πολύ τοξικό όταν συσσωρεύεται και ιδιαίτερα επιζήμιο για την ανθρώπινη υγεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να στηρίζουμε συνεχώ όλα τα συστήματα διαλογή, συλλογή και ανακύκλωση, προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε μια ανακύκλωση τη τάξη του 100% όσον αφορά τι τεχνικέ στήλε και του ερευτές που χρησιμοποιούν κάδμιο. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, ε, τεχνολογίες αντικατάστασης. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε για παράδειγμα στήλες ιόντων λιθίου, οι οποίες είναι βέβαια πιο ακριβές και ενδεχομένως να μην ιδιαίτερα δημοφιλείς στις πιο φτωχές χώρες. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαγορεύσει μέχρι το 2015 τη χρησιμοποίηση καδμίου είναι προφανώς ένα διοικητικό μέτρο που υποστηρίζει κάποιες νέες τεχνολογίες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι νέες αυτές τεχνολογίες είναι πιο ακριβές. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί ένας καλύτερος συμβασμός που να λαμβάνει υπόψη και τις οικονομικές δυνατότητες των Ευρωπαίων πολιτών. Ενδεχομένω να έπρεπε να έχουμε ως 2016 καταληκτική ημερομηνία απαγόρευσης ή ακόμα και αργότερα. Σας ευχαριστώ ο κύριος Μίρσκι για ένα μισή λεπτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Διάβασα πάρα πολύ προσωπικά την πρόταση του κύριου Παναγιώτοφ Είμαστε πολύ καλοί φίλοι με τον κύριο Παναγιώτοφ. Χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερα να συνεργαστώ μαζί του πάρα πολύ επικοδομητικά για τη σημαντικότατη αυτή έκθεση. Η έκθεση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσουμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων από τις πολύ αρνητικέ επιπτώσεις του υδραργίου, υδραργύρου και άλλων τοξικών βαρέων μετάλλων. Πολύ συχνά επικρίνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο σήμερα θα ήθελα να χαιρετήσω την πρόταση αυτή. Βλέπουμε ότι έχει γίνει μια επαγγελματική δουλειά και βλέπουμε ότι και οι επιπτώσει αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ θετικέ. Ξέρετε ότι το κάδμιο είναι ένα πολύ επικίνδυνο μέταλλο, το ίδιο ισχύει και για τον υδράργυρο και η απαγόρευση των βαρέων αυτών μετάλλων προφανώ θα διασφαλίσει ένα υψηλότερο επίπεδο υγεία για όλου του Ευρωπαίου πολίτε. Και οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι θα δουν επίση ότι εμεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργαζόμαστε πολύ καλά. Βλάτκο, πραγματικά είμαι πάρα πολύ περήφανο για την δουλειά που έχει κάνει και χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργαστήκαμε πάρα πολύ επικοδομητικά. Και εξ ονόματο πολιτική μου ομάδα πρέπει να πω ότι στηρίζουμε την κοινή αυτή εργασία που έγινε με τον κύριο Παναγιώτοφ και με την συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Περάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Μέσαρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο Παναγιώτο αυτόν εισηγητή μας, για την ε, εξαιρετική του έκθεση. 40% όλων των ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων, όλων των ηλεκτρικών εργαλείων ε, είναι ασύρματα με βάση τις περσινές ε, στατιστικές. Και τα περισσότερα από τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούν ηλεκτρικές στήλες νικελίου καδμίου που, είναι, που ξαναφορτίζονται. 70% είναι των λιθίου και 20 λιθίου και άλλων μετάλλων. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη όμως ότι στην Ανατολική Ευρώπη οι αναλογίες είναι ανάποδες. Έχουμε πολύ περισσότερες ε, στήλες νικελίου και θα χρειαστούμε πολύ περισσότερο χρόνο και μεταβατική περίοδο για να απαγορεύσουμε τέτοιες ουσίες, ε, την χρήση καδμίου δηλαδή σε τέτοιες ηλεκτρικές στήλες. Σίγουρα ε, το κάδμιο είναι πολύ τοξική ουσία και δεν ξέρουμε πόσο καιρό χρειάζεται για την ε, απεικοδόμησή του. Θα πρέπει λοιπόν όμως να δούμε πώς θα ανακυκλώνουμε τις ηλεκτρικές στήλες ε, που περιέχουν κάδμιο. Σίγουρα θα βρούμε μια ρεαλιστική λύση που θα εξυπηρετήσει και τις βιομηχανίες αλλά και τους καταναλωτές. Ευχαριστώ. Ο κύριος ακόμα προϊόντα που περιέχουν ε, κάδμιο κυκλοφορούν. Ε, κυρίως ε, μπαταρίες, ε, ιατρικά προϊόντα. Είναι μια πάρα πολύ τεξική, τοξική ουσία το κάδμιο για το περιβάλλον και για τον άνθρωπο. Πρέπει λοιπόν να αντικατασταθεί με άλλες όπως παραδείγματος χάρη το λίθιο. Το θέμα δεν αφορά μόνο τις μπαταρίες, ακόμα και λιπάσματα στη μη βιολογική καλλιέργεια περιέχουν κάδμιο. Οπότε σχεδόν σε κάθε τρόφιμο υπάρχει αυτή η τοξική ουσία. Πρέπει λοιπόν να φύγει όχι μόνο από τις ηλεκτρικές συσκευέ, αλλά και από τα τρόφιμα. Και πρέπει να υποστηρίξουμε τη σχετική έρευνα για την ε, έβρεση αναλλακτικών και βεβαίως να ενισχύσουμε τα βιολογικά προϊόντα. Σας ευχαριστώ. Ε, κυρία Μαγκίνης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζω πως έχουμε επισκέπτες στο Κοινοβούλιο και ο τίτλος συζήτησης είναι βαρετός. Αλλά η ουσία είναι πάρα πολύ σημαντική και για τους επισκέπτες και τους πολίτες μας. Ξέρω πως ο Φιλ Χόγκαν από την Ιρλανδική Προεδρία είχε παίξει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη συμφωνίας ε, που δίνει μια βεβαιότητα και στην βιομηχανία αλλά και στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία για το ότι τα βαρέα αυτά και τοξικά μέταλλα θα απαλληφθούν από τις μπαταρίες. Ε, χτες λοιπόν είχα μια ομάδα επισκεπτών και ήταν ενδιαφέρον ε, να ακούσω τις απόψεις τους για την Ευρώπη και ανέφερα πως ε, όταν μιλάμε για τη διάθεση των αποβλήτων, αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ιρλανδία δεν θα είχαν συμβεί χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις οδηγίες της. Και αυτή είναι εδώ. Και τα πράγματα γίνονται αργά. Αλλά όταν λαμβάνει αποφάσεις η Ευρώπη, τα αποτελέσματα είναι ορατά και είναι πάντα προς το όφελος της δημόσιας υγείας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Και βεβαίως τον λόγο τώρα έχει και ο κύριος Κέλλη μια που ακούσαμε για την Ιρλανδική Προεδρία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους ιδιαίτερα στον εισηγητή, όχι μόνο για το αξιόλογο έργο του στον πολύ σημαντικό αυτό τομέα, που μπορεί να μείνει το πιο σεξι θέμα στον κόσμο, το πιο ελκυστικό, αλλά σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα ήθελα όμως να τον ευχαριστήσω για τις πολύ καλές ε, και ε, πρακτικές διευκρινήσεις που μας έκανε για το έργο που έχει γίνει, δίνοντας έμφαση στην ε, ανάγκη για μια ανώδυνη μετάβαση, την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, αλλά και ταυτόχρονα είπε ότι πέντε τόνοι υδραργύρου εκλείονται στο περιβάλλον κάθε χρόνο. Σίγουρα θα πρέπει κάπως να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Χάρη όμως στο δικό του έργο και στο έργο της Επιτροπής θα έχουμε μια βελτίωση. Και οι δύο εμπειρογνώμονε συνάδελφοι πίσω από μένα μίλησαν για τα σύρματα ηλεκτρικά εργαλεία και την ανάγκη να βελτιώσουμε την, ε, ε, τον τρόπο κατασκευή ε, κατασκευής και τα υλικά που χρησιμοποιούν. Πολύ σημαντικό όμω είναι και το θέμα της ανακύκλωσης γιατί μερικές ηλεκτρικές στήλες απλώς απαιτιούνται από τον κόσμο γιατί δεν ε, υπάρχει αρκετή συνειδητοποίηση. Ενώ ξέρουν ότι πρέπει να ανακυκλώνουν ε, πλαστικά, αλουμίνιο, χαρτί, δεν γνωρίζει ο κόσμος ότι πρέπει να ανακυκλώνουν και τις μπαταρίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο Επίτροπος Ευκόντς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καλείστε να εγκρίνετε μια αναθεώρηση επικαιροποίηση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις ηλεκτρικές στήλες και τους ισορρευτές. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και καταφέρνουμε να διευκρινίσουμε κάποιες σημαντικές διατάξεις στις οδηγίες προκειμένου αυτή να εφαρμοστεί καλύτερα. Όπως είπε λοιπόν η κυρία Μαγκίνες, αφού είναι πάρα πολύ καλό για τους πολίτες, για την υγεία τους, είναι καλό για το περιβάλλον και θεωρώ ότι ε, παρέχει την απαραίτητη ε, σαφήνεια και διαφάνεια για τους επιχειρηματίες. Σας ευχαριστώ πολύ που στηρίζετε λοιπόν την πρόταση αυτή οδηγίας. Να απαντήσω τώρα σε ένα ερώτημα που έθεσε ο κύριος Σλίτερ. Θα ήθελα να τον διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται το ζήτημα το οποίο έθιξε αντιμετωπίσουμε κάποιες τεχνικές δυσκολίες με την ομοιόμορφη σήμανση, ιδίω για τις ηλεκτρικές στήλες οι οποίες δεν επαναφορτίζονται. Πάντως συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με διάφορους οργανισμούς τυποποίησης και συγκεκριμένα και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης, το ΣΕΝ, ο οποίος μας βοηθά να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για να επιλύσουμε το ζήτημα αυτό. Μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να έχουμε μία σήμανση κατά περίπτωση, αλλά βέβαια επεξεργαζόμαστε το ζήτημα το οποίο θίξατε και προφανώς θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε πρόοδο σημειώσουμε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο εισηγητής, ο κύριος Παναγιώτοφ. Okay. Тъй като съм развълнуван, ще говоря на родния си български язик. Благодаря, господин президент, господин комисар, уважаеми колеги. Тази директива и изказванията по нея. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω βεβαίω στην ε, γλώσσα μου. Σα ευχαριστώ λοιπόν για τα καλά σα λόγια και αυτό το οποίο άκουσα σήμερα ε, και η δουλειά βεβαίω με τους συναδέλφους ε, κατέδειξαν πως ε, πράγματι μπορούμε να κάνουμε κάποια σημαντικά πράγματα εδώ και χρόνια μιλάμε για ένα αποτέλεσμα και τελικά καταλήξαμε φέτος σε έναν συμβιβασμό συμβιβασμό στον οποίο συμφωνούν Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Κομισιόν και έτσι βεβαίως καταφέραμε σε κάτι το οποίο αφορά ιδιαίτερα τις χώρες που έχουν ε, λιγότερη αγοραστική δύναμη. Είμαι απολύτως ε, σίγουρος ε, πως θα βοηθήσουμε έτσι και την τεχνολογική εξέλιξη της Ευρώπης χωρίς ε, τους ε, σκιώδεις ε, εισηγητές, χωρίς τους συναδέλφους που συνεισέφεραν σε αυτό το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή. Και εδώ πέρα τελειώνει αυτό το θέμα. Η ψηφοφορία σήμερα στις 12 η ώρα. Θα λέμε σε λίγο. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, διακόπτεται η συνεδρίαση.